αξιότιμοι συνάδελφοι κυρίες και κύριοι επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης καθώς και τα εγκεκριμένα κείμενα ε, διατίθενται. Έχετε διαφωνίες, αντιρρήσεις, όχι. Οπότε και θεωρούνται εγκεκριμένα τα συνοπτικά πρακτικά. Και